ο κύριος Χάν. Uh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίε και κύριοι, μας ε, προκάλεσε φρίκη οι εικόνες ε, των νεκρών τουριστών στην παραλία της Τίνιδας. Πρόκειται για μια επίθεση που ήθελε να σπείρει φόβο στεκόμαστε μαζί με τους ίσιους για να αποτύχουν οι τρομοκράτες. Ήταν μια επίθεση ενάντια σε ανθρώπους. οι Τα συλληπιτήριά μας πηγαίνουν με τις στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλο τον λαό της Τινησίας. Ήταν μια επίθεση στην θαραλέα επιλογή της Τινησίας υπέρ της δημοκρατίας. Χτύπησε τον τουρισμό, ζωτική, ζωτικό κλάδο της οικονομίας της χώρας ενώ η χώρα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Η δημοκρατική μετάβαση της Τινησίας από το 2011 και μετά είναι μοναδική. Θεωρείται και από τους ίδιους τους ε, Τινήσιους αποτέλεσμα της ε, ιστορίας τους, αλλά παραμένουν πολλές προκλήσεις για τη χώρα. Χρειάζονται πολλές θαραλέες μεταρρυθμίσεις για να παγιωθεί το, συνταγμα, το δημοκρατικό σύνταγμα της χώρας και να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες της χώρας που επηρεάζουν κατά βάση την νεολαία της χώρας. Η Ένωση υποστήριξε τις προσπάθειες της χώρας αυτής από το 2011 και θα συνεχίσει να το κάνει ε, καθώς η κυβερνή είναι ε, βασική, ε, βασικός προορισμός των εξαγωγών της χώρας. Εμείς προτείνουμε την επένδυση στη χώρα αυτή. Είναι κοινή ευθύνη μας να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν με ασφάλεια. Οι επιθέσεις δεν ήταν το πρώτο δείγμα των τεράστιων προκλήσεων της ημισίας. Μετά την Επανάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ε, συνεργαστεί με τις αρχές της χώρας ένα διάλογο για μια συνολική μεταρρύθμιση του τμήματος του χώρας, του, της ασφάλειας στη χώρα ούτως ώστε τα όργανα ασφάλειας να μπορούν να παράσχουν καλύτερη ασφάλεια στους πολίτες με σεβασμό των διεθνών ε, κανόνων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εξασφαλίζουν που εξασφαλίζει το νέο σύνταγμα. Παρά τις δυσκολίες ε, που είναι εγγενείς σε τέτοια αναπτυξιακά προγράμματα τόσο μεγάλου μεγέθους, το πρόγραμμα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή που έχει δεσμευθεί να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις, μας επιτρέπει να βοηθήσουμε σημαντικά. Θα επιταχύνουμε όσο περισσότερο γίνεται την εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Σαν τμήμα των ε, μεταρρυθμίσεων θα δώσουμε έμφαση στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης ε, των πολιτών της χώρας στα όργανα ασφάλειας. Ωστόσο θέλουμε να υπογραμμίσουμε ακόμα περισσότερο μαζί με τον συντονιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης για να βρούμε ευκαιρίες άμεσης δράσης με όλα τα εργαλεία που υπάρχουν για να βοηθήσουμε την, την, την Ισία να διαμορφώσει την αντιτρομοκρατική στρατηγική της, ιδίω την αντιμετώπιση της ρίζοσπαστικοποίησης και την ενίσχυση των μηχανισμών ασφάλειας. Η κυρία Μογκερίνη έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό της Ισία τον Μάιο με μια σειρά συγκεκριμένων προτάσεων. Και εγώ έγραψα στον Υπουργό Ανάπτυξης Επενδύσεων και Διεθνούς Εμπορίου της Ισία αμέσως μετά την επίθεση στη Σούσα για να τον διαβεβαιώσω ότι η Ένωση στηρίζει σταθερά την, την Ισία και ότι θα επιταχύνουμε την ε, μεταφορά κάποιων ε, δόσεων της ενίσχυσης που κανονικά θα πήγαιναν αργότερα φέτος. Το παράδειγμα της Τινησίας δείχνει ότι οι τρομοκράτες επιτίθεται στην Ισία γιατί είναι επιτυχία. Είναι μια επιτυχής προσπάθεια εκδημοκρατισμού. Καλό την Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη να υποστηρίξει την χώρα αυτή με μια πλουραλιστική δημοκρατική κυβέρνηση και μια κοινωνία που θέλει να προστατεύσει την, τα δικαιώματα των γυναικών και τα ατομικά δικαιώματα. Πρέπει να υπάρχει κινητοποίηση όλων των πόρων που είναι διαθέσιμα ε, σε εμά για να υποστηρίξουμε τη μετάβαση της χώρας προς τη δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση που θα αποδεικνύουν την κοινή αποφασιστικότητά μας. Επίσης, η επιχειρησιακή βοήθεια είναι σημαντική. 187 εκατομμύρια ευρώ σε διμερή βοήθεια μόνο για το 2015. Ωστόσο, προτίθεμαι να διερευνήσω κάθε δρόμο για να ενισχύσω περαιτέρω την προσπάθεια αυτή η μακροοικονομική βοήθεια είναι ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να αυξηθεί τα επόμενα έτη. Τούτου λεχθέντος βεβαίως η χώρα είναι μια χώρα σε εξαιρετικά σταθή περιοχή. Η προστιθέμενη αξία είναι ανάλογη με το μέγεθος της χώρας και την κρίσιμη περίοδο της αλλαγή των αλλαγών που υφίσταται η χώρα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η συνεισφορά μας θα παράσχει, θα απορροφηθεί σωστά γιατί το να δίνουμε χρήματα δεν λύνει την κατάσταση. Η υποστήριξη στην Τινησία είναι στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και αυτό απαιτεί και ταχύτητα και ευελιξία σε κάποιες περιπτώσεις. Ταυτόχρονα ωστόσο απαιτεί και προγραμματισμό. Η Τινησία ήταν ο κύριος δικαιούχος των λεγόμενων ταμείων ομπρέλα που παρέχουν ε, χρηματοδότηση σε συγκεκριμένους επιλεγμένους εταίρους που προωθούν τη δημοκρατία φέτος, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες της νησίας για την εφαρμογή των στόχων αυτών, προτείνουμε ένα επιπρόσθετο ποσό γύρω στα 70 εκατομμύρια ευρώ <coughs> για να αντιμετωπίσουμε τις θετικέ εξελίξεις. Μετά τα πρόσφατα γεγονότα εξετάζουμε βέβαια και πώς θα βελτιώσουμε καλύτερα τις προσπάθειες να ενισχύσουμε τις προτεραιότητες μας αυτές. Πολλά μένουν να γίνουν για να παγιώσουμε την ε, νέα δημοκρατία της Ινησίας Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ασφάλειας ε, ε, είναι καθοριστικές. Η μετάβαση απαιτεί να υπάρξουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, να υπάρξει ένα ευνοϊκό κλίμα για ανάπτυξη και επενδύσεις. Ε, πρέπει να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι προκλήσεις με προσπάθειες πολλών ετών και σε όλους τους τομείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να προσφέρει βοήθεια στην Τινησία. Επίσης μπορούμε να διαδραματίσουμε καθοριστικό ρόλο ε, στο να εμπλουτίσουμε την προνομιούχο εταιρική σχέση που έχουμε με την Τινησία. Η Τινησία ε, βεβαίω ε, μπορεί να υποφεληθεί από τις κοινοτικέ πολιτικές. Αυτές προσφέρουν περαιτέρω ευκαιρίες στις ε, εταιρικές, στις χώρες, στους εταίρους μας. Παραδείγματο χάρη, ανταλλαγές σε επίπεδο πανεπιστημίων, στην έρευνα, στην καινοτομία, στη γεωργία, καθοριστική σημασία τομέα για τη χώρα. μαζί με τους συναδέλφους μου θα αναζητήσουμε τις δυνατότητες για επιπρόσθετες δράσεις. Θα δώσουμε σημασία σε πράξεις που θα οδηγήσουν στη δημιουργία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 την αγανάκτησή μου στο Σούσα αλλά και στο Μουσείο Μπάντεν να εκφράσω τα βαθιά μου συλληπιτήρια στους οικείους των θυμάτων. Νομίζω λοιπόν έχουμε κάθε λόγο να στηρίξουμε αυτή τη νεόκοπη δημοκρατία, να τη στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Εγώ προσωπικά ήδη το 2011 πήγα επί τόπου ως ε, Chief Observer, κύριος παρατηρητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ήμουνα και στις δεύτερες εκλογές μαζί με συναδέλφους. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι οι Τινήσοι επιθυμούν αυτή τη δημοκρατία. Σε αυτές τις εκλογές δεν εμφανίστηκαν ακραίοι, παρότι ε, το όριο για να μπει κανείς στο κοινοβούλιο ήταν πολύ χαμηλό. Οι Τινήσοι όμως δεν θέλουν εξτρεμισμό και γι' αυτό πρέπει να τους στηρίξουν στηρίξουμε στις προσπάθειές τους. δείξατε και εσείς ορισμένα στοιχεία. Για μένα είναι σημαντικό να ελέγξουμε ένα επιπρόσθετο στοιχείο και παρακαλώ αυτό να το συζητήσετε με την κυρία Μογκερίνη. Όπως γνωρίζετε υπάρχει ε, μια αποστολή, μια συνεργασία μεταξύ την Ισίας ε, και Λιβύης. Αυτή έχει ανασταλεί, ε, περιμένει να δει καλύτερες ημέρες. Κατά την άποψή μου θα ήταν σημαντικό να ελέγξουμε το κατά πόσον μπορούμε να έχουμε μια αποστολή Ευρωπαϊκής Ένωσης CSDP επιτόπου με τους ε, Τινήσιους έτσι ώστε να παρεμποδίσουμε την ε, διείσδυση τρομοκρατών και άλλων παρεμφετών τρών στοιχείων. Γιατί ο ε, τρομοκράτης και στο Μουσείο και στο Ζούζι εκπαιδεύτηκε εκεί στη Λιβύη. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το προσφέρουμε ως συγκεκριμένη βοήθεια και θα ήθελα να ελέγξετε κατά πόσο αυτό είναι δυνατό. Για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών το λόγο έχει ο κύριος Τζάνι Πιτέλα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, συνάδελφοι, Εξ ονόματος της ομάδας μου θέλω να εκφράσω τα βαθιά μου συλληπιτήρια προς τις οικογένειες, την κυβέρνηση και το λαό της Τινησίας ε, για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. Επιθέσεων που θέλουν να καταστρέψουν την ιδιωτική μάχη των ε, Τινήσεων για αξιοπρέπεια και ελευθερία. Θέλουν να μετατρέψουν την Τινησία που δεν θέλουν να μείνει η Τινησία το μόνο καλύτερο παράδειγμα της ε, ε, Αραβικής Άνοιξης. Θέλουν να κάνουν αυτό το παράδειγμα ένα τρομοκρατικό κράτος. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Δεν αξίζει στο λαό της Τινησίας. Πρέπει να προστατεύσουμε την σταθερότητα της, της δημοκρατίας της χώρας και να διευκολύνουμε την μετάβαση προς μια δημοκρατία. Γι' αυτό λέω προς εσάς κύριε Πίτροπη και προς την κυρία Μογκερίνη να αναλάβετε μια ισχυρή πολιτική, θεσμική και ηθική δέσμευση να είστε στην πρώτη γραμμή εσείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο με βάση την θέση σας αλλά και με συγκεκριμένες προτάσεις να προτείνουμε ένα πρόγραμμα Marshall για την, ε, την Ισία, γιατί επλήγει σε ένα νευραλγικό τομέα της ε, οικονομίας της, τον τουρισμό, που είναι βασικό συστατικό της οικονομίας της. Χρειάζεται λοιπόν συγκεκριμένη βοήθεια, γιατί αυτό είναι το βασικό στοιχείο των σχέσεων Ένωσης και Μεσογείου. Είναι ένα στοιχείο βασικό για τη μετάβαση στη δημοκρατία της κοινωνίας αυτής. Δεν μπορούμε να πούμε όχι στην στρατηγική προοπτική μας για την, Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή Συνεργασία. Αυτό είναι το νόημα των πρώτων πρόγραμμα Μάρσαλ. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ζητούν από εσά και από την κυρία Μογκερίνη να αναλάβετε δράση σε, αυτό το, σε αυτή τη σημαντική πρόταση για αυτή τη μεγάλη υλοποίηση. Λεπτό για την ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών ο κύριος Τάνοκ. Uh, Πρόεδρε, η τρομοκρατική επίδεση στην Τινησία ε, ε, δημιούργησε απώλεια 39 ζωών μεταξύ των οποίων και Βρετανών πολιτών ίσως και της περιφέρειάς μου και ε, εκφράζω τα συλληπιτήριά μου σε όλους τους φίλους και τις συγγενείς τους. Και άλλες φορές έχουν γίνει τέτοιες επιθέσεις κοντά στο Μουσείο Μπάρντο στην Τίνιδα. Η Τινησία χρειάζεται ζωτικά την λήψη μέτρων. Ήταν από τις χώρες που είχαν πρωταγωνιστήσει στην Αραβική Άνοιξη και η πτώση της δικτατορίας του Μπεναλή άνοιξε το δρόμο για την πολυκομματική δυτικού τύπου δημοκρατία. Τώρα η κυβέρνηση του Χαμπίμπεψη ίσως επιτρέψει στην Τινησία να ανθίσει ως ένα σύγχρονο κράτος κοσμικού χαρακτήρα. Το 10% του ΑΕΠ της Τινησίας αντιπροσωπεύεται από τον τουρισμό και γι' αυτό είναι τρομερή ζημία η επίθεση αυτή. Και η λήψη μέτρων θα ήταν σημαντική για το μέλλον της χώρας. Ευχαριστώ. Την ομάδα Φιλελευθέρων και Δημοκρατών το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Ντεσαρνέζ. Ε, Επίτροπε, όλοι το ίδιο λέμε. Φυσικό είναι. Οι τρομοκράτες χτύπησαν δύο φορές σε τρεις μήνες στην Ισία, στην Πάρντο και στην Τσούση. Αυτό είναι αυτό γιατί η νέα η νεαρή δημοκρατία στην Ισία πάει καλά. Γιατί η μετάβαση προς τη δημοκρατία πάει καλύτερα. Και γι' αυτό θέλουν να πλήξουν οι τρομοκράτες. Άρα προφανώς απαιτεί να είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση δίπλα στους Τινήσιους, δίπλα στην Τινησία. Πρέπει να είμαστε παρόντες ε, και στο επίπεδο ασφάλειας, στη διαχείριση του ελέγχου των συνόρων με τη Λιβύη, για παράδειγμα, κάτι προφανές πρέπει να είμαστε παρόντες στο θέμα των μεταναστευτικών ροών, να διαχειριστούμε μαζί τους το, τις ροές μεταναστών και την ίση και Ευρωπαίης και πρέπει να είμαστε παρόντες οικονομικά. Μιλήσατε για την ε, αποστολή, ταχύ αποστολή χρημάτων. Πρέπει να βοηθήσουμε ωστόσο να υπάρξουν βιώσιμα προγράμματα που θα κρατήσουν χρονικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτή οι επενδύσει να είναι προ όφελο της Τινησίας διαφυλάσσοντας ε, τομεί που είναι ζωτικοί για αυτήν, υπηρεσίες, ε, γεωργία και η Ευρώπη πρέπει να δώσει το παρόν, μιλώντας, ε, όντας δίπλα στην Τινησία, δίπλα στους Τινήσιους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Προομάδα της αριστεράς, το λόγο έχει η κυρία Βερζιά για 1,5 λεπτό. Monsieur le Président. Η φρίκη χτύπησε ξανά τρεις μήνες μετά την Πάρκο στην Ισία, στο Σούσα. Και εγώ να στείλω τα συλληπιτήριά μου στη χώρα αυτή, μια μικρή χώρα, 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπου ο τουρισμός, ο τουρισμός είναι πραγματικός πνεύμονας οικονομικός. Η Τιμησία εκεί ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη και είναι, Άνοιξη και είναι η μόνη χώρα που συνεχίζει την ε, πορεία προς τη δημοκρατία. Οι τρομοκράτες γι' αυτό χτύπησαν εκεί. Η αλληλεγγύη μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Αυτό δεν συμβαίνει ωστόσο. Η Τινησία χρειάζεται ε, βοήθεια στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά δεν θα πρέπει να τεθούν επαμφιβόλω τα, τα μικρά κέρδη της δημοκρατίας μετά την Επανάσταση και να έχει μια οικονομική ανάπτυξη που θα δώσει προοπτική στην νεολαία. Μέχρι τώρα η Ισία έλαβε πολύ λίγα. Ακόμα και από την βοήθεια που χρησιμοποιήθηκε κατά βάση ως υπομορφή ε, δανείων που επιδίνωσαν την, ε, την υποχρέωση, τη χρέωσή της. Τα σύνορα με την Ευρώπη μένουν κλειστά. Πρέπει να Κύριε Πίτροπε, είστε εδώ για να ακούσετε. Άρα ακούτε αν γίνεται. Εντάξει. Λέω ότι είναι καιρό, να σταθούμε στο ύψο μας, θέτοντα νέο πλαίσιο συνεργασία, αντιμετωπίζοντας το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέου και ένα μορατόριο ενδεχομένω, ενισχύοντα την περιφερειακή συνεργασία προ όφελο των φτωχότερων χωρών με πραγματική εταιρική σχέση προ όφελο του λαού τη χώρα οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να καθοδηγηθούν μόνο με μεγαλύτερη απελευθέρωση προς όφελος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε την Τινησία. Είναι επίγον και πρέπει να γίνει προτεραιότητα. Πολιτική ομάδα των Πρασίνων, ο κύριος Σεμπαστιά για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με την ευκαιρία θέλω να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου προς τα θύματα των, της επίθεσης στην Τίνιδα. Πριν λίγους μήνες είχα, ήμουν παρατηρητής ε, για το κοινοβούλιο στην Τίνιδα ενώπιση των εκλογών και μαζί με κάποιους συναδέλφους εδώ και είδα ότι η διαδικασία ήταν ελεύθερη, διάφανη και γεμάτη ελπίδα. Η αποστολή είχε πολλές συναντήσεις με πολλούς εκπροσώπους, πολιτικούς, υποψήφιους, κοινωνία των πολιτών, τον τωρινό πρόεδρο μεταξύ άλλων, που θύμισαν ότι η Αραβική Άνοιξη ήταν ένα σύνολο διαφορετικών συνθήκων. Η πραγματική άνοιξη ήταν η Τινήσια άνοιξη, η μόνη χώρα όπου υπήρξε δημοκρατική ρήξη με επιτυχία. Ταυτόχρονα μας έλεγαν ωστόσο πιο διακριτικά ότι οι νήσοι αισθάνονταν μόνοι, Μόνη μέσα σε μια περιοχή γεμάτη συγκρούσεις με πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Λιβύη και τρομοκράτες. Τι έκανε μέχρι τώρα η Ευρώπη. Τα χρήματα που έδωσε για την Τίνιδα είναι, ε, ανέρχονται σε γελίο ποσό. Όλα, όλοι απαιτούν την υποστήριξή μας. Στον τομέα της ασφάλειας είναι σαφές. Σε πολιτικό είναι σαφές, αλλά κυρίως οικονομική βοήθεια χρειάζεται για να έχει μια σταθερότητα και να μπορέσει η νεολαία, ένας χώρος που πλήττεται ιδιαίτερα, που, ελκύεται κυρίως από τους δημοκράτες πρέπει να ενισχυθεί. Σε αυτό το, το σύνολο του νότου της Μεσογείου πρέπει να βλέπουμε λίγο περισσότερο από ό,τι βλέπαμε. Προ, επίτροπε χρειαζόμαστε σαφή δέσμευση έναντι της πόλης γιατί ε, αυτό, ε, από αυτό εξαρτάται η δική μας για ομάδα Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Καστάλντο. Ευχαριστώ, Πρεσιδέντε 21 νεκροί στο Πάντο, 31 στο Πόρτα Αλκατάου στην Σούσα. Κατάσταση εκτακτου ανάγκη στην χώρα. Ο στόχο των τρομοκράτων είναι προφανώ να καταρρεύσει ο τουρισμό, ένα κλάδο βασικός τη οικονομία. Η χώρα από αυτό ζει. Γιατί αυτή η λύσα ο λόγο είναι απλός. Η Τινησία είναι ένα ούνικουμ στον αραβικό κόσμο, η μόνη πραγματική δημοκρατική μεταπολίτευση που υπάρχει, που γίνεται. Με δυσκολία αλλά που γίνεται. Ε, με ένα ε, χώρο σταθερότητα. Αυτή η αλλαγή τρομοκρατεί πολλού, του τρομοκράτε, αλλά και κάποια αυταρχικά αραβικά καθεστώτα που δείχνουν σαφώ την συμβατότητα μεταξύ Ισλάμ και Δημοκρατία. Πάντα είναι ε, ανάρμοστο κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ενοχλεί η Τινησία. Η Τινησία ωστόσο είναι πολλές Τινησίες. Είναι το κομμάτι των ακτών που είναι πιο δυτικό, πιο τουριστικό, πιο παραγωγικό. Που και αυτού η περιοχή πλήττεται από μια ανεργία. Υπάρχει η ενδοχώρα που είναι φτωχή, που είναι ο βασικός πυρήνας των foreign fighters. τρει με τέσσερι χιλιάδες. Ζήτησα στην Επιτροπή ΑΦΕΤ να υπάρξει μια ειδική έκθεση για τη χώρα αυτό. Πιστεύω ότι η αξία αυτής της έκθεσης πηγαίνει πολύ μεγα... είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος της χώρας και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Σπιτέλα όταν έλεγε ότι χρειαζόμαστε ένα σχέδιο Μάρσαλ. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε τομείς τόσο σημαντικούς όπως ε, η ασφάλεια ή θέματα μετακυκλικής μετανάστευσης. Πρέπει να περάσουμε ένα κοινωνικό ευρύ πρόγραμμα. Η εμπειρία μας είναι μια προσπάθεια να μειώσουμε το, το χρέος. Αλλιώς αν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα στεκόμαστε στο ύψος της χώρας αυτής. Αν το κάνουμε αυτό θα έχουμε ένα ακραίο καθεστώς το οποίο μπορεί να πάρει το Μαγκρέμπ ολόκληρο μαζί του. Ο λαός της Τινησίας έχει την υποχρέωση να αντιμετωπίσει καλύτερα την κατάσταση. Είναι, όλοι το ζητούμε αυτό διότι οι, πιστεύουν στη δημοκρατία και αν σπάσουν τις αλυσίδες αυτό θα εξαρτηθεί και από εμά. Ας μην του αφήσουμε μόνους, μόνους τους. της το λόγο έχει για 1,5 λεπτό κύριος Merci, euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά σκεφτόμαστε όλοι τα θύματα των επιθέσεων στην Τινησία. Θα ήθελα να χαιρετήσω εδώ την απόφαση του Τινήσιου Προέδρου ΕΣΕΠΣΥ που κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και έθελε να κλείσει πολλά σαλαφιστικά τζαμιά. Κατά τα άλλα, το δίκαιο που είχε αρχίσει να εφαρμόζει ο Μπουργκίμπα και συνέχισε ο Μπέναλι συνεχίζει να εφαρμόζεται. Τελευταία στις 18 Μαρτίου και στις 26 Ιουνίου σημειώθηκαν αυτές οι επιθέσεις και υπόθηκε ότι στη Δινησία υπάρχει ο μεγαλύτερος αριθμός ριζοσπαστικών μουσουλμάνων. Στην Αλγερία υπάρχουν επίσης τρομοκρατικά κομμάντο όπως και στη Λιβύη. Στην Τινησία από το 2012 οι τρομοκράτες ε, έχουν ανεβεί στο βουνό και όλα αυτά δεν μας δείχνουν τίποτε το καλό. Το κόμμα Εναχντά θεωρείται εναλλακτική λύση. Είναι Ισλαμιστικό μεν κόμμα αλλά περιμένει την ευκαιρία του. Από τον περασμένο Οκτώβριο μπόρεσα να συναντήσω πολιτικούς της Τινησίας και εκεί έμαθα ότι η Εναχντά καραδοκεί και μπορεί να οργανωθεί με το πρότυπο των αδελφών μουσουλμάνων της Αιγύπτου. Δυστυχώς οι Ευρωπαίοι πολιτικοί δεν έδειξαν καμία φρόνηση για να αντιμετωπίσουν την απειλή αυτή. Το κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω προσθέτοντας ε, και τη δική μου την αίσθηση αλληλεγγύης και κατανόησης ε, προς τον λαό της Τινησίας. Εκφράζω τα θερμά μου ε, συλληπιτήρια στις οικογένειες ε, των ε, θυμάτων αυτών των τραγικών τρομοκρατικών επιθέσεων. Η Τινησία είναι το καλύτερο παράδειγμα για δημοκρατική μετάβαση της Αραβικής Άνοιξης. Υπάρχουν βέβαια εκείνοι που ενδιαφέρονται να αποσταθεροποιήσουν την Τινησία και θέλουν να αποδείξουν ότι το Ισλάμ είναι συμβατό με τη δημοκρατία. Η Τινησία χρειάζεται πηγόντως την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιτύχει το στόχο της σταθερότητας, πολύ περισσότερο μάλιστα σήμερα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαν ως στόχο τους ε, τουρίστες για να υπονομεύσουν τον τουρισμό σε μια περίοδο εχμής. Χρειάζονται λοιπόν ουσιαστική, οικονομική και ε, τεχνική βοήθεια και το ε, θέλω να πω, το λέω ε, σε απόλυτη συμφωνία με τον κύριο Πιτέλα, ο οποίος μίλησε για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την Τινησία. Το να βοηθήσει κανείς την Τινησία σημαίνει επίσης ότι θα βοηθηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν υπάρχει μια σταθερή δημοκρατική χώρα, αυτό θα είναι το καλύτερο παράδειγμα για το τι μπορούν να επιτύχουν και να επιδιώξουν οι χώρες της ε, περιοχής. Έχουν ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις η χώρα έχει νέο σύνταγμα. Ε, εδώ λοιπόν απευθύνομαι σε εσά, ε, κύριε επίτροπε, και στην υπατή εκπρόσωπο να βοηθήσετε στην υλικοτεχνική υποδομή ε, να υπάρχουν πληροφορίες για τους τρομοκράτες και η Τινησία θα πρέπει να μπορεί να απευθυνθεί καλύτερα στους Ευρωπαίους. Το λόγο έχει η κυρία Σάικε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι, όπως κάθε λογικός άνθρωπος και εγώ σοκαρίστηκα από την δειλή επίθεση των τρομοκρατών σε την Ισία και εκφράζοντας λυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων. Αυτό μας θυμίζει όμως ότι η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική δεν μπορούν πάντα να αποσυνδεθούν. Παρά τη λύπη μας για τις τρομερές αυτές επιθέσεις δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η Τινησία είναι και ε, μια ε, μεγάλη επιτυχία μετάβασης από τη δικτατορία σε μια ανοιχτή κοινωνία. Οι Τινήσιοι πριν από πέντε χρόνια βγήκαν στους δρόμους ζητώντας μια πιο δίκαια και δημοκρατική κοινωνία. Η μετάβαση βέβαια δεν είναι ποτέ εύκολη αλλά πολλοί νέοι που είχαν βαρεθεί πλέον την ε, διαπλοκή και τη διαφθορά. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το ξεχάσουμε τα αιτήματα αυτά δηλαδή. Θέλουμε η Τινησία να παραμείνει ένας βασικός εταίρος μας και να τη βοηθήσουμε να οικοδομήσει μία διαφοροποιημένη και δημοκρατική ανοιχτή κοινωνία. Το τελείως αντίθετο δηλαδή του μηδενιστικού δόγματος του πολιτικού Ισλάμ που δρά μόνο μέσω της βίας. Προσωπικά δεν θα ήθελα να σκέφτομαι με όρους βοήθειας προς την Τινησία αλλά συνεργασίας με την Τινησία και οι ανακοινώσεις διαπραγματεύσεων για εμπορικές συμφωνίες συμφωνούν με αυτή την αντίληψη για να δημιουργηθεί μια πιο ελεύθερη κοινωνία με ευκαιρίες για όλους τους Τινήσιους ιδιαίτερα τους νεότερους. Έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος ναι, ευχαριστώ. Πέραν των συλληπιτήριων που πρέπει να δώσουμε, εμεί πρέπει να πούμε ότι η επίθεση στο ΣΟΥΣ, η δεύτερη μέσα σε δύο μήνες, είχε ένα αποτέλεσμα, ότι τέθηκε σε ισχύ η κατάσταση εκτά του ανάγκης. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι αναγκαία, αλλά δείχνει τα προβλήματα που υπάρχουν ένα πλαίσιο ανασφάλεια στη χώρα που μπορεί να αποσταθεροποιήσει σοβαρά την, το μέλλον της χώρας. Δεύτερον, το, ότι ο κίνδυνος ε, να μειωθούν τα πολιτικά δικαιώματα λόγω του, της κατάστασης ανάγκης, κάτι αρνητικό για την παγίωση της μεταπολίτευσης και της δημοκρατίας. Στην κατάσταση αυτή χρειαζόμαστε να υπάρξει μια δέσμευση, ουσιαστική δέσμευση ενίσχυσης της δημοκρατίας, ιδίως διότι η χώρα, χώρα αυτή πρέπει να προχωρήσει προς την αντιμετώπιση της δημοκρατίας και τη σταθερότητα. Ο ρόλος της Ευρώπης είναι καθοριστικός. Το είπαμε σε πολλά ψηφίσματά μας. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Χρειάζεται να υπάρξει μια πιο σωστή προσέγγιση στην, για την Ινσία. Μιλήσατε, Επίτροπε, για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα Δυστυχώς δεν είμαστε φιλόδοξοι προς το παρόν. Χρειάζεται μία, ε, μία βοήθεια παρόμοια με αυτή που δώσαμε στην Ουκρανία και αν θέλουμε να βοηθήσουμε πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. Η θεσμική και δημοκρατική στερέωση του πειράματος της χώρας είναι κάτι από το οποίο εξαρτάται και η ασφάλεια της περιοχής και η δική μας. Ευχαριστώ, Presidente. Primero, mis condolencias a las víctimas. Και εγώ να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προς τα θύματα των επιθέσεων. Πρέπει να πούμε τι γίνεται σε μια χώρα που έχει την θρησκευτική πολιτιστική και πολιτιστική παράδοση της χώρας τόσο ώστε ένας νέος μηχανικός να γίνει τζιχαριστής. Τι γίνεται με τη ματέωση τόσων πολλών νέων στη χώρα αυτή. Είναι προφανές ότι η στρατηγική ασφάλεια είναι κλειδί, αλλά δεν είναι το μόνο κλειδί και δεν είναι αρκετό. Αν δεν αναπτυχθεί η Τινησία, δεν μπορούμε να παγιώσουμε την δημοκρατική διαδικασία. Και για να υπάρξει ανάπτυξη χρειαζόμαστε περισσότερο από του Κοινοβουλίου ή μικρά προγράμματα χρηματοδότησης. Αν θέλουμε να υπάρξει μια δημοκρατία στις πύλες της Ευρώπης που μπορεί να θριαμβεύσει που να είναι το μόνο θριαμβευτικό αποτέλεσμα των αραβικών ανοίξεων χρειαζόμαστε να δουλέψουμε πραγματικά και δεν το κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, μας είπε ο, μας πρόεδρος όταν είχαμε πάει στην Τινησία τότε ότι ένα, ένα, ένα χελιδόνι δεν φαίνει την άνοιξη. Που έχει για Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ακόμη μια φορά έχει υποστεί τρομοκρατία η Τινησία με τις επιθέσεις αυτές που ακόμη μια φορά την πλήττουν. Πρέπει λοιπόν να επαναλάβουμε το μήνυμα αλληλεγγύης μας προς τους Τινήσιους και τις Τινήσιες. Και ταυτόχρονα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα για να στηρίξουμε τον εταίρο μας αυτόν. Νομίζω κύριε Επίτροπε ότι πρέπει καταρχάς να επιτρέψουμε στον Ομπάμ Λίμπια να επιστρέψει για να μην γίνει η Τινησία μόνο ένα μαξιλάρι μεταξύ Αλγερίας και Λιβύης. Έπειτα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε ακόμη περισσότερο όπως είπε και ο συνάδελφος Παντζέρη την Τινησία και στη νέα μας ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας να προσπαθήσουμε η χρηματοδότηση αυτή να είναι πιο σημαντική. Αυτοί είναι οι δύο άξονες που πρέπει να ακολουθήσουμε κύριε Επίτροπε, ώστε επιτέλους να μπορέσουμε να επιδείξουμε πραγματική αλληλεγγύη στην πράξη με την Τινησία. Που έχει για ένα λεπτό Η στην ε, Αφρική καταβάλλονται προσπάθειες ε, να καταπνιγεί η δημοκρατία που προέκυψε στην Τινησία. Είχαμε λοιπόν επιθέσεις σε παραλίες, σκοτώθηκε ένας Πορτογάλος, άρα η τρομοκρατία δεν γνωρίζει ε, σύνορα. Οι τρομοκράτες συνεργάζονται και προσιλητίζουν ανθρώπους λόγω της ανεργίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν με την πολιτική της ε, συνέβαλε να εξελιχθεί αυτή η πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει την ευθύνη να καταπολεμήσει το Ισλαμικό κράτος και ε, σε εμά, στη Λιβύη και στην Τινησία πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, πρέπει να στηρίξουμε τις δημοκρατικές εξελίξεις μιας χώρας ε, έτσι ώστε να υπάρξει κάποιο μέλλον για τους ε, νέους σε αυτή τη χώρα. Να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία, άρα δηλαδή πρέπει να υπάρχουν ασφαλείς δρόμοι για μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Ε, όχι να επιτρέπουμε ε, τη δραστηριοποίηση των ε, διακινητών. Γιατί αλλιώ θα έχουμε επιθέσεις και στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν πρέπει να στηρίξουμε την Τινησία, να στηρίξουμε το δημοκρατικό έλεγχο σε αυτή τη χώρα. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Γκίλ. Και εγώ καταδικάζω τις τρομερές επιθέσεις στην Τινησία που στόχευσαν κυρίως Ευρωπαίους πολίτες Πολλοί ήταν Βρετανοί και μερικοί και από τη δική μου περιφέρεια των West Midlands. Αυτό μας θύμισε τις προηγούμενες επιθέσεις που είχαμε υποστεί και θα ήθελα να εκφράσω λοιπόν και εγώ τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. καθώς και σε όλους τους ανθρώπους που είδαν τη χώρα τους να υφίσταται επίθεση για δεύτερη φορά σε λίγους μήνες. Η Τινησία είναι παράδειγμα για πολλές χώρες και γι' αυτό υπόδειγμα και γι' αυτό πρέπει να τη βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο για να διασφαλίσουμε ότι η κατάσταση πολιορκίας που θα χρειαστεί να επιβληθεί θα συμφοβαδίζει παρόλα αυτά με τα πρότυπα του διεθνούς δικαίου. Επειδή ο τουρισμός είναι η, ο δεύτερος η δεύτερη πλουτοπαραγωγική πηγή της Τινησίας, τα μέτρα ασφαλείας για αυτόν τον τομέα είναι ζωτικά και για το μέλλον της Τινησίας. Λεπτό, η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Gracias, presidente. Sí, mi solidaridad y simpatía en primer lugar para todo Túnez, pero también para las familias de las víctimas, ciudadanos europeos, cierto, pero también. Είμαστε πολίτες της Τινησίας ενώπιον της επίθεσης στον Πάντο όπως και στο Σούσα όπου είδαμε εικόνες Τινήσιων που προστατεύουν τις, ε, με, τη, ζωή τους τους Ευρωπαίους τουρίστες γιατί έχουν επίγνωση ο τουρισμός, ότι ο τουρισμός είναι πηγή πλούτου για αυτούς. Δεν έχουν πετρέλαιο όπως οι γείτονες και το ξέρουν αυτό διότι και οι τρομοκράτες διότι χτύπησαν στην Τίνιδα, το μόνο, στο Τίνιδα, το μόνο, τη μόνη πηγή πλούτου της μόνης δημοκρατίας στην αραβική χώρα. Την πιο ειρηνική χώρα της περιοχής. Μας, ε, το ότι χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν κατά την τζιχάντα, άνθρωποι αυτοί που, το, που την άνοιξη του, το χειμώνα και την άνοιξη του 2010 αγωνίστηκαν για να κάνουν δημοκρατία την ε, χώρα τους. Τι κάναμε εμείς όλο αυτόν τον καιρό σε Ευρωπαίοι, τίποτα σε σχέση με άλλες περιοχές που βοηθάμε μαζικά. Στην Τίνιδα, ε, στο Νότο βρίσκεται η ασφάλειά μας, η βασική μας ασφάλεια, η ανάγκη τόσων νέων να, να γίνει κάτι για τη δημοκρατία και το μέλλον τους. Γι' αυτό ζητούμε ένα πρόγραμμα που ζήτησε η χώρα και που ακόμα περιμένουμε, Επίτροπε. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών. Προχωρούμε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχω δεχτεί τρία αιτήματα, αλλά από ό,τι βλέπω ο κύριος Φρουντζουλίτσα δεν είναι τώρα παρόν. Επομένως προχωράμε στους δύο παρόντες. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η τελευταία τρομοκρατική επίθεση στην Τινησία συγκλώνησε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και ιδίως το Βέλγιο και τη Γαλλία. Ταυτόχρονα είχαμε όμως και την ε, απόφαση να τεθεί η τινησία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το οποίο ε, δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα για τη δημοκρατική πορεία της χώρας αυτής. η ευρωπαϊκή ένωση είναι σίγουρο ότι πρέπει να έχει μια στρατηγική για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας των τζιχαντιστών και η πρώτη παρέμβαση που πρέπει να κάνει η ευρωπαϊκή ένωση αφορά την οικονομική ανάπτυξη της τινησίας να χτυπηθούν δηλαδή οι οικονομικές και οι κοινωνικές αιτίες που έχουν προκαλέσει τη φτώχεια και την υπανάπτυξη στην περιοχή αυτό για να γίνει πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του εξωτερικού χρέους της τινησίας. τον θυμόσαστε κύριοι συνάδελφοι τον περίφημο δικτάτορα της τινησίας τον μπεν αλή που επί 23 χρόνια κυβερνούσε την τινησία που ήταν το αγαπημένο παιδί του δουνουτού που όταν έπεσε από την εξουσία βρέθηκαν εκατομμύρια ευρώ στο σπίτι του επομένως το βασικό θέμα είναι να υπάρξει διαγραφή του εξωτερικού χρέους της τινησίας προς το δελτα τη γαλλία την ιταλία και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Γιάκοφτσης. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Nije slučajno izabran Κύριε Πρόεδρε. napad. I naravno nije slučajno izabran η Τινησία δεν επελέγει κατά τύχη. Και συμπτωματικά πλήγει και η τρομοκρατία και ο τουρισμός από αυτή την τρομοκρατική πράξη. Είχαμε πολλούς αθώους, πάρα πολλές οικογένειες και βεβαίως εμείς επιθυμούμε να τους εκφράσουμε τα συλληπιτηριά μας και σε όλους τους πολίτες. Κύριε Επίτροπε, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε ειρήνη και ασφάλεια σε αυτή την περιοχή και αυτό προϋποθέτει διάφορες μορφές βοήθειας, καταρχήν θεσμική βοήθεια και μέτρα ασφάλειας. Όμως πρέπει να κάνουμε περισσότερα διότι την Ισία είναι μια χώρα που μπορεί να αποτελέσει μοντέλο ε, για άλλες χώρες που έχουν προβλήματα μετά την Αραβική Άνοιξη. Η Τινησία είναι ένα καλό παράδειγμα. Ας διαφυλάξουμε λοιπόν τη χώρα όσο μπορούμε. της Αντιπροέδρου της Επιτροπής κυρίας Μογκερίνη, ο Επίτροπος κύριος Χάν. Κύριε Χάν, έχετε το λόγο. Vielen Dank, Präsident. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους ε, όσοι έλαβαν ε, το λόγο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, διαβεβαιώσω ότι η νησία είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας και δεν χρειαζόταν να λάβουν χώρα αυτές οι τραγικές τρομοκρατικές επιθέσεις και ούμονον αυτό αλλά πρότεινα στην κυβέρνηση της Τινησίας ε, να τους βοηθήσουμε όχι μόνο για να δείξω την αλληλεγγύη μας αλλά και για να πείσω τους Ευρωπαίους πολίτες ότι πρέπει να πάνε στην Τινησία να περάσουν εκεί τις ε, διακοπές τους μου είπαν ότι αυτή τη στιγμή καλύτερα να μην πάω γιατί έχουν πάρα πολλά και άλλα προβλήματα πάντως ε, πρέπει να δείξουμε ότι τους στηρίζουμε ε, συμμερίζομαι και αυτά που είπατε σχετικά ε, με το πρόγραμμα Marshall. Πράγματι δεν πρόκειται μόνο για την Τινησία, πρόκειται και για άλλες ε, χώρες της περιοχής και αυτές οι χώρες θα ήταν δυνάμει υποψήφιες χώρες ε, αποδέκτες ε, ενός προγράμμου, προγράμματος Marshall του 21ου αιώνα. Η Παγκόσμια Τράπεζα διαθέτει τεχνογνωσία και γι' αυτό πιστεύω και εγώ ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε, να βοηθήσουμε μόλις προσφερθεί η ευκαιρία. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι στην Τενησία έχουμε ε, ουσιαστική παρουσία και σήμερα το βράδυ θα μας δοθεί η δυνατότητα ε, στο πλαίσιο της έκθεσης Κούκαν να μιλήσουμε για την αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας. Ο πρωταρχικός μας λοιπόν στόχος και νομίζω επ' αυτού συμφωνούμε όλοι είναι να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα στην περιοχή για να το πετύχουμε όμως αυτό από την άλλη πλευρά πρέπει να επιδείξουμε και ευελιξία για να μπορούμε να αντιδράσουμε και θα ήθελα λοιπόν ήδη τώρα να σας ε, παρακαλέσω οποτεδήποτε χρειαστούμε την ευελιξία ε, για να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα να μας στηρίξετε κι εσείς. Τα θέματα της ασφάλειας, οι σχετικές προτάσεις που κατατέθηκαν θα τα λάβω ιδιαίτερα υπόψη μου. Ξέρω ότι είπα ότι εκπρόσωπος ε, έχει δραστηριοποιηθεί για αυτά τα θέματα ε, και βεβαίως αναζητά τις δυνατότητες που υπάρχουν για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και σε σχέση με τη Λιβύη. Και τέλος ε, θέλω να σας πω ότι η Τινησία θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη ε, του επόμενου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών στις 20 Ιουλίου. Έχουμε καλέσει τον Ταϊπακούς, τον Υπουργό Εξωτερικών της Τινησίας, να μας κάνει ε, την παρουσία τους κατά τη διάρκεια του γεύματος, γιατί εκεί γίνονται περισσότερες άτυπες συζητήσεις. Η συζήτηση έληξε. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής υπά της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής